Αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια... Πρώτο θέμα στην ημερήσια... Α, συγγνώμη, κύριε Σασόλη, θέλετε το λόγο. Point of order, παρακαλώ. Όχι, ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε και σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Χθε το βράδυ οι αστυνομικέ δυνάμει στην Ιταλία συνέλαβαν πέντε άτομα τα οποία προετοίμαζαν μια μαφιόζικη επίθεση κατά του συναδέλφου Ροζάριο Κροτσέτα, μέλο του Κοινοβουλίου και πρώην δημάρχου μία πόλη στη Σικελία, τη Τζέλα. Σύμφωνα με του δικαστέ, από σήμερα ε, στι 20 του Ιανουαρίου ε, ε, θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε στιγμή για την οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσε να γίνει η απόπειρα αυτή. Θα πρέπει να δούμε το θέμα της προστασία του συναδέλφου, ο οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς στην Ιταλία, όπω γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε. Καλώ την Προεδρία λοιπόν να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον συνάδελφο να εκφράσει λοιπόν η Ολομέλεια την αλληλεγγύη της ε, προς ε, τον συνάδελφο και να ε, λάβουμε κάθε μέτρο έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματική προστασία του κυρίου Κροτσέτα κατά την ανάπτυξη των καθηκόντων του ως μέλος του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ θερμά κύριε Σασόλη. Είχατε απόλυτο δίκιο να θέσετε το ζήτημα αυτό στην Ολομέλεια. Ε, σας ευχαριστώ. Πρώτο θέμα στη μερίσια διάταξη είναι η εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή υπό το άρθρο 204 του κανονισμού. Έχω λάβει τρεις υποψηφιότητες με αλφαβητική σειρά. Ο κύριος Βιτόριο Μποτόλη, ο κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος και ο κύριος Pierre Μονέτ. Οι υποψήφοι πρέπει να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία των ψηφισάντων και υπό αυτό το πρίσμα οι αποχές δεν προσμετρώνται. Γυρνώ τώρα στα αγγλικά γιατί πρέπει να κάνουμε ένα τεστ. we will have to start a brief test. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαδικασία ελέγχου δοκιμής για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τουλάχιστον 368 μέλη εδώ στην αίθουσα όπως ορίζεται από τον κανονισμό, το ξέρω, το ξέρω, αλλά θα το ελέγξουμε. Και θα σας αρέσει γιατί θα είναι πολύ επίμαχη η ψηφοφορία. Να επαναλάβω τις οδηγίες, τις οποίες τις έχετε μπροστά σας, στις γλώσσες σας. Καταρχάς, Καταρχάς θα πρέπει να τοποθετήσετε τον Κέρσορα στο όνομα του υποψηφίου που θα ψηφίσετε και αυτό θα γίνει με τα δύο μπλε κουμπιά που έχετε στα δεξιά και να πιέσετε μετά το πλήκτρο συν και μετά θα ανάψει ένα μπλε φωτάκι όχι πράσινο, όχι πορτοκαλί, μπλε για όλους και θα εμφανιστεί μπροστά από το όνομα του υποψηφίου. Ωραία ως εδώ. Ωραία. Αν θέλετε να δηλώσετε ότι συμμετέχετε χωρίς να ψηφίσετε, θα, πατήσετε το 0. Τρίτον, μπορείτε να αλλάξετε την ψήφο σας πρωτού ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, επανεπιλέγοντας τον πρώτο υποψήφιο και πατώντας το 0 και μετά περνώντας με τον κέρσορα στον δεύτερο υποψήφιο που θέλετε πραγματικά να ψηφίσετε και να πατήσετε το συν επειδή είναι πολύπλοκη η διαδικασία, θα κάνουμε έναν έλεγχο, μία δοκιμή. Έχουμε λοιπόν τους τρεις ε, υποψήφιους με αλφαβητική σειρά. Θα ελέγξουμε και μάλλον θα τεθεί σε κρίση και το πολιτισμικό και η πολιτισμική κρίση του Κοινοβουλίου Πικάσο, Ρενουάρ και Βαγκόγκ. Εντάξει λοιπόν, έτοιμοι έναρξη ψηφοφορία. Okay, everyone should vote. Να ψηφίσετε παρακαλώ όλοι. Μετακινήστε τον κέρσορα στο όνομα της επιλογής σας. Πατήστε το ανάλογο κουμπί. <laughs> Okay. Has, has everyone... El Greco, they didn't ask me, Mr. Τον Αλγκρέκο δεν τον έχουμε βάλει. Δεν με είχαν ρωτήσει, αλλιώ θα τον είχα προτείνει. Ψήφισατε λοιπόν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. The vote is closed. Okay. Πέρας ψηφοφορίας ήταν πολύ οριακό το αποτέλεσμα. 240 ψήφι Van Gogh, Renoir 238 και 166 ψήφοι για τον ε, Πικάσο. what would have the majority been here? Okay, now, I think we're ready. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να περάσουμε στην ψηφοφορία. Να περάσουμε το νέο κατάλογο. Με το ίδιο σύστημα ακριβώ θα ψηφίσουμε. Χειροκροτάτε για το Bangkok ή τι θέλετε το λόγο. Συγγνώμη, αλλά δεν λειτουργεί το δικό μου μηχάνημα, κύριε Πρόεδρε. Σα το συγγνώμη, αλλά δεν λειτουργεί. να I don't have... Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. It Φαίνεται ότι ο κύριος Van ε, θέλει και αυτός να υποβάλει υποψηφιότητα για διαμεσολαβητής, γιατί δεν βγαίνει από τη λίστα. Προσπαθούμε να τον αλλάξουμε. Είμαστε έτοιμοι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Θα δείτε τα ονόματα στην οθόνη σας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. συγκέντρωσαν ο κύριος Διαμαντούρος 340 ψήφους από τους 678, ο κύριος Μονέτ 289 ψήφους, ο κύριος Μποτόλη 19 ψήφους. Έχουμε λοιπόν την επικράτηση του κυρίου Διαμαντούρου από την πρώτη ψηφοφορία Συγχαρητήρια στον κύριο Διαμαντούρο και αν θέλει μπορεί να, ε, να βγει παρακαλώ. Ε? Και συγχαρητήρια και σε όλους τους άλλους υποψηφίους. Πέρασαν από μια πολύ δύσκολη διαδικασία ακροάσεων και στην Επιτροπή και στις πολιτικές ομάδες και ήταν και οι τρεις ε, αξιολογότατοι συγχαρητήρια σε όλους. Είναι εδώ ο κύριος Διαμαντούρος. On behalf of the On behalf of the Commission, the floor is to Commissioner Wallström. Δίνουμε το λόγο στην Επίτροπο Thank you very much, Mr. President, honorable members. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και αξιότιμα Αξιότιμοι βουλευτέ, να συγχαρώ τον Δικήφορο Διαμαντούρο που εξελέγει στη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Όπω αναφέρθηκε στην έκθεση του, του περσινού έτου, το βασικό του καθήκον είναι η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι συμμεριζόμαστε το στόχο αυτό και θα πρέπει να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση και είναι σημαντικό καθήκον αυτό και για το θεσμού μας αλλά και για εμάς ως άτομα. Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διαμεσολαβητή ήταν πάντα πάρα πολύ καλές και πολύ επικοδομητικές. Η συνεργασία μας θεωρώ ότι έχει καταστεί ακόμα πιο ομαλή και αποδοτική και μέσα από τις έρευνές τους ο διαμεσολαβητής έχει βοηθήσει πολύ στην ε, ανάπτυξη μιας ατμόσφαιρας εξυπηρέτησης ε, του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέπουμε ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη προθυμία για την επίτευξη φιλικών διακανονισμών. Θα πρέπει να συνεχιστούν αυτές οι εξελίξεις και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες του διαμεσολαβητή και θα καλωσορίζει πάντα τις ε, προτάσεις του. Τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ ε, δύσκολα αλλά και ενδιαφέροντα για τον ε, Ευρωπαίο διαμεσολαβητή χάρη και στις νέες δυνατότητες που δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Η καλή διακυβέρνηση, όπως ξέρετε, αναφέρεται ρητά στον χάρτη των θεμελιδών δικαιωμάτων. Δεν ε, αμφιβάλλω ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για να ενισχύσει την δημοκρατία, τη διαφάνεια και τους θεσμούς προς όφελος του πολίτη. Όλοι έχουμε ευθύνη να συνδράμουμε στο έργο του αυτού. Και πάλι λοιπόν σας συγχαίρω για το διορισμό σας και φυσικά σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τα σημαντικό καθήκον που έχετε μπροστά σας. πολύ την κυρία Βάλστρομ και την ε, Επιτροπή. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία επί της ε, εκθέσεως της κυρίας Χούμπνερ σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζόρων. Σας επισημαίνω ότι υπάρχει ένα διορθωτικό το οποίο αφορά όλες τις γλωσσικές αποδόσεις της έκθεσης αυτής. Τη θέτω σε μοναδική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Σβανγκό. Είμαστε έτοιμοι νομίζω. Άρχεται η ψηφοφορία. Επιτρέψτε μου τότε στο ενδιάμεσο να πω στον κύριο Διαμαντούρο uh, that I hereby invite you to swear the oath before the Court of Justice in accordance Σας καλώ λοιπόν να προχωρήσετε στην, στο ενορκομοσία με βάση ενώπιον του ε, δικαστηρίου σύμφωνα με τους ε, κανόνες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 628 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια στην κυρία Χούπνερ. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία τη πρόταση απόφασης, σχετικά με την πρόταση διορισμού της Άννα Παλάσιο ε, Βαλαρεσούντι στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Τέλος. Τέλος, η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία από τις έκθεσης της ε, κυρίας ε, Τζολί σχετικά με τη δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Συμφωνία του Κοτονού Και περνάμε στις τροπολογίες. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 496 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται με 397 ψήφους υπέρ. Σας παρακαλώ, ναι, έχετε το λόγο. Uh, we send uh, τροπολογία 3. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. εγκρίνεται με 392 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 4 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 509 ψήφους υπέρ, Herr Schulz. Dankeschön. Dankeschön for the help. Uh, τροπολογία 5 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με 300, 304 ψήφους κατά και πάμε τώρα στην τελική ψήφο επί του συνολικού ψηφίσματος ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά Αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Τζολή. Και περνάμε τώρα στις ε, αιτιολογήσεις ψήφου. Πρώτα για την ε, εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ο κύριος Μπονσινιόρε. Con questo voto il Parlamento με την ψήφο αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο